Συνεχίζουμε. Κοινή συζήτηση για την νομιμοποίηση εισόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ε, σύσταση για δεύτερη ε, ανάγνωση με συνεισηγητές ε, τους Κιγιάννης Κάριντσε και Ζούντις Σαργεντίνη. Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση τρομοκρατίας. Έχουμε αυτή την σύσταση για δεύτερη ανάγνωση, καθώς επίσης και μια άλλη σύσταση πάλι για δεύτερη ανάγνωση, τον Τίμωθη Κίρκοπ και Πίτερ Σάιμον. Τον ε, κύριο Κάρεν καλό πρώτα να πάρει τον λόγο. Εκ των συνεισηγητών. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι, σήμερα και αύριο θα ολοκληρωθεί η διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια. Έχουμε αναπτύξει νέα νομοθεσία για να καταπολεμήσουμε το ξέπλυμα χρήματος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σαρτζεντίνη, την συνεισηγήτρια, τους συναδέλφους από την Επιτροπή ΛΥΜΕ και την ε, Ιταλική Προεδρία γιατί καταλήξαμε σε συμφωνία επί Ιταλικής Προεδρίας. Τι πετύχαμε λοιπόν τα δύο αυτά χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να βελτιωθεί η νομοθεσία για την καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος. Και οι προτάσεις της Κομισιόν εγκρίθηκαν, δηλαδή ότι θα γίνεται μια προσέγγιση με βάση την αξιολόγηση κινδύνου και έτσι θα μπορούν οι τράπεζες να μαθαίνουν κάποια πράγματα παραπάνω για τους πελάτες τους και θα υπάρχει μια μαύρη λίστα η οποία θα βοηθάει τις διοκτικές αρχές και το τραπεζικό τομέα να έχουν περισσότερες πληροφορίες για τους πελάτες τους όσον αφορά δε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε προτείνει ένα νέο μέσο το οποίο μας βοηθά να βρούμε μία άκρη, δηλαδή το ευρωπαϊκό μητρό του πραγματικού ιδιοκτήτη. Μέχρι τώρα έχουμε διάφορα εμπορικά μητρό και τέτοια άλλα. Βεβαίως οι ιδιοκτήτες μπορούν να είναι ιδιώτες ε, φυσικά και νομικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα είναι η ιδιοκτησία άλλων νομικών προσώπων κτλ. κτλ. και δημιουργούνται αλυσίδες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και κανείς δεν ξέρει ποιος είναι πίσω από μια συγκεκριμένη εταιρεία. Η πρότασή μας, η οποία υπάρχει και στην ε, πρόταση αυτή της νομοθεσίας, είναι πως θα υπάρχει μια απέτηση σε όλα τα κράτη-μέλη να υπάρχει ένα μητρό του ε, πραγματικού ιδιοκτήτη. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα έχουμε τώρα αυτή την αλυσίδα υπεράκτιων εταιριών που δυσκολεύει τις ιδιοκτικές αρχές και θα μπορούμε επιτέλους να αποκαλύψουμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης πίσω από μια εταιρεία και μια συναλλαγή. Και αυτό θα βοηθήσει και στη συλλογή των φόρων. Γιατί αυτά χρησιμοποιούνται όχι μόνο για το ξέπλυμα αλλά και για την ε, φοροδιαφυγή. Νέα εξέλιξη λοιπόν έχουμε τώρα η οποία θα αναγκάσει τους ε, εγκληματίες να αντιδράσουν. Και βεβαίω θα κάνει όλα αυτά τα συστήματα να δυσκολευτούν πάρα πολύ. Στην Ευρώπη έχουμε κράτος δικαίου, έχουμε κάποια συστήματα τραπεζικά και χρηματοδότησης και με την αλλαγή της νομοθεσίας. θα γίνει πιο αποτελεσματική η καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος και θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και θα πάει σε τρίτες χώρες. Σας ευχαριστώ λοιπόν και παρακαλώ αύριο να υπερψηφίσετε το σχέδιο αυτό. Σας ευχαριστώ κύριε Κάρινς. Θα δώσω τώρα τον λόγο στην κυρία Σαρτζεντίνη για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ και τον κύριο Κάρινσε, τον συνεισηγητή μου και τους ε, σκιώδης που βοήθησαν και σε αυτή την περίοδο αλλά και την προηγούμενη περίοδο. Επίσης τον Ρομπέρτο Κροτσέρη από την ε, πρόεδρο της Επιτροπής, Γουαλτιέρη, ε, της Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν πολύ μακρά η διαδικασία αυτή. Ξεκινήσαμε στην προηγούμενη θητεία και καταφέραμε να τελειώσουμε το προηγούμενο Δεκέμβρη και να σας πω ότι είχαμε και μία ε, ψηφοφορία στην Ολομέλεια ε, στην προηγούμενη ε, θητεία που έδωσε στον κύριο Κάρινς μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία 603 υπερψηφισάντων για την δημιουργία του ενός μητρώου. Αυτά όλα έγιναν έχοντας σαν κύριο μέλημα ε, την φοροαπαλλαγή και την φοροδιαφυγή. Είναι τεράστια τα ποσά ε, τα οποία φεύγουν ε, από την Αφρική. Το ακούσαμε επανειλημμένα εδώ στο σώμα γιατί οι πολυεθνικές δεν πληρώνουν φόρους. Είναι σκανδαλώδηση η κατάσταση. Επίσης για την περίπτωση της Ουκρανίας που έκλεψε χρήματα χρήματα στην ουσία από, τον Ουκρανικό λαό για να τα βάλει σε τράπεζες ε, της ε, Ολλανδίας ε, και είχαμε και το LuxLeaks τελικά το οποίο μας έδωσε όλες αυτές τις πληροφορίες για τα tax rulings. Ultimate beneficial owners. εν πάση περιπτώσει, εμείς συμφωνήσαμε να έχουμε 28 αρχεία ε, και ε, τώρα οι χώρες οι οποίες δεν είχαν μέχρι τώρα πρέπει να δημιουργήσουν αυτά τα μητρώα. Τα μητρώα όμως θα είναι ε, διασυνδεδεμένα και θα έχουν την δυνατότητα να ελέγχουν αναχώρα και ανα επιχείρηση, αναεταιρεία. Φυσικά οι δημόσιες αρχές είναι αυτές οι οποίες μπορούν να ελέγχουν τις εταιρείε, επιχειρήσει, τα καζίνο κτλ. Αλλά και όσοι έχουν ένομο συμφέρον θα μπορούν ε, να το κάνουν αυτό και να ελέγχουν. Γιατί υπάρχουν θέματα παρανόμων δραστηριοτήτων, νομιμοποίηση εσόδων, χρηματοδότηση τη τρομοκρατία κτλ. Οι δημοσιογράφοι και οι μη κυβερνητικέ οργανώσει επίση και ο κάθε ε, μεμονωμένο πολίτη μπορεί να ε, ε, ελέγξει τα μητρώα αυτά έτσι ώστε να σταματήσει πλέον αυτή η δυνατότητα που έχουν οι εταιρείε να κλέβουν λεφτά από τους φόρους ε, και να τα κλέβουν από την κοινωνία, από την δημόσια εκπαίδευση, από την υγεία κτλ. Και εμείς θέλουμε να πάμε ακόμα παραπέρα, να είμαστε βεβαίως και προσεκτικοί. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ρόφα γιατί μόλις ε, ε, άρχισε να ασχολείται με τα θέματα αυτά, κάναμε ένα βήμα προόδου όσον αφορά την προστασία ε, των προσωπικών δεδομένων, γιατί πρέπει να είναι σαφές ότι ο καθένας ο οποίος θεωρεί ότι με κακό τρόπο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα του θα πρέπει να έχει δυνατότητα δράσης. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα σβηστούν οποιασδήποτε εγκληματικές δραστηριότητες ή θα προστατεύσουμε εγκληματίες. Κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτό ε, να αποτελέσει ένα παράδειγμα για άλλες χώρες του κόσμου. Δεν θα ήταν καταπληκτικό εάν μας ακολουθούσαν ε, και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, θα θέλαμε να, σας, να μας βοηθήσετε έτσι ώστε στον τομέα της φοροαπαλλαγής και της φοροδιαφυγής να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κέρκοφ τώρα για τέσσερα λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, εάν δεν έχουμε ροή χρημάτων προς ε, τους ε, τρομοκράτες, τότε καταπολεμά κανείς και το ξέπλυμα και την τρομοκρατία. Το πρόβλημα που δημιουργεί η νομοποίηση παρανόμων εσόδων είναι τεράστιο και βεβαίως η διαφάνεια είναι ένα πολύ ισχυρό όπλο. Έχουμε μία ευκαιρία που εμείς χρησιμοποιήσαμε μαζί με τους συνεισήγητες και τους σκιώδες και για το θέμα αυτό πρέπει να σου πω πως αισθάνομαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος. Εξετάσαμε ποια είναι τα διεθνή πρότυπα και το γεγονός πως πρέπει το θέμα αυτό να το αντιμετωπίσουμε και πέραν των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα υπόλοιπα κράτη του κόσμου. Θα πρέπει να μπορούμε να παρακολουθούμε τη δρομή του χρήματος σε άλλες χώρες, να μπορούμε να κατασχέσουμε ε, περιουσία και να μειώσουμε την ε, ευελιξία κινήσεων των ε, εγκληματιών. Με τον τρόπο αυτό θα παρακολουθήσουμε τη διαδρομή του χρήματος πέρα από τα δικά μας σύνορα. Εδώ και πολλά χρόνια έχουν οι προσπάθειες οι οποίες δεν ήταν πετυχημένες. Ο στόχος μας ήταν τούτη τη φορά να έχουμε μία αναλογική, λογική και αποτελεσματική λύση που θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε στη μάχη κατά της νομοποίησης του παράνομου χρήματος. Ε, πρέπει να σας πω πως τελικά η νομοθεσία την οποία είχαμε προωθήσει εδώ στο ε, παρελθόν ε, ίσχυσε στο Ηνωμένο Βασίλειο με έναν τρόπο που έκανε τη, τη ζωή δύσκολη στους μικροεπενδυτές ε, χωρίς ουσιαστικά να φέρει αποτελέσματα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να επαναλάβουμε τέτοιου είδους προσπάθειες ε, άσκοπα. Θα πρέπει να δούμε ποιε θα είναι οι επιπτώσει στην ιδιωτική ζωή και πώς θα προστατεύσουμε τα ιδιωτικά δεδομένα. Αυτό το λάβαμε δεόντως υπόψη. Αναλογικότητα και αναγκαιότητα είναι όροι που χρησιμοποιούμε συνέχεια στις προσπάθειες που κάνουμε στο Κοινοβούλιο και νομίζω ότι εδώ είναι ακόμα πιο σημαντικέ αυτέ οι λέξει. Στο παρελθόν πολλέ φορέ δόθηκαν κάποιες ε, δυνατότητες ε, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να χρησιμοποιήσουν τρόπους ε, πολύ επιτακτικούς και περιγραφικούς για να αξιολογήσουν τις πελάτες τους. Όχι, θα πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να αξιολογούν τους πελάτες τους με ένα αξιόπιστο σύστημα αναφοράς και όχι απλώς να υπογράφουν ε, τα κράτη-μέλη τα διεθνή πρότυπα, αλλά να εξασφαλίζουν και την αγαστή συνεργασία με τρίτες χώρες για να επενδύουν οι εταίροι μας από τις άλλες χώρες στην Ευρώπη και για να μεγαλώσει η ευρωπαϊκή αγορά χρειαζόμαστε κατάλληλα νομικά εργαλεία, ευρωπαϊκή συνεργασία για να προλαμβάνουμε και να διώκουμε το οικονομικό έγκλημα. Ελπίζω αυτό το οποίο παραδίδουμε να είναι εύχριστο, να λειτουργήσει και για μένα η δυνατότητα του να εφαρμοστεί αυτό το πακέτο ήταν και η πρώτη ε, ανησυχία η οποία με καθοδήγησε γιατί όσο καλή και να είναι η νόμη σου αν δεν εφαρμοστούν στην πράξη δεν κερδίζεις κάτι και πιστεύω πως με το πακέτο αυτό θα αποκομίσουμε μεγάλα κέρδη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους συνεισέφεραν και τον κύριο Σάιμονς Σκιώδη τους άλλους ε, συνεισηγητές και τους υπόλοιπους σκιώδες συνεισηγητές και ελπίζω η αυριανή ψηφοφορία να αποτελέσει μια αφετηρία στη μάχη κατά του ξεπλήματος χρήματος έτσι ώστε να υπάρξει και αποδοχή σε επίπεδο κοινή γνώμης για τις προτάσεις που υποβάλαμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κέρχοφ. Ο Πίτερ Σίμον είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκτιμάται πως ε, 1.600 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο ξεπλένονται. 3% του παγκοσμίου ΑΕΠ. Μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή είναι ένα τρισεκατομμύριο κάθε χρόνο. Ένα ποσό μεγαλύτερο από το επταετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωση. Εμείς, άρα ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το ξέπλυμα χρήματο όπω και την ε, φοροδιαφυγή. Εξού λοιπόν ε, και η επεξεργασία της τρίτης οδηγίας ε, του 2005. Οι σοσιαλδημοκράτες όσον αφορά την τρίτη αυτή οδηγία, την τέταρτη οδηγία της Κομισιόν την υποστηρίζαμε πάντα και, τα, και τον σχετικό κανονισμό και οι δύο, τα δύο αυτά νομοθετήματα προτείνουν μια προσέγγιση η οποία βασίζεται στην αξιολόγηση κινδύνου. Δηλαδή θα εστιαστούμε σε κλάδους που έχουν υψηλό τέτοιο κίνδυνο για ξέπλυμα χρήματο. Και ακριβώς αυτό φαίνεται και στο πεδίο εφαρμογής. Στο μέλλον θα δούμε και τα καζίνα και ε, τους παρόχους τυχερών παιγνίων. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι, κατά την άποψή μας, και η διαφάνεια και άρα το να διαπιστώνουμε ποιος ε, είναι ο πραγματικός ε, ιδιοκτήτης ε, πάρα πολλών εταιρικών κατασκευών και εταιριών γραμματοκιβωτίων. Γι' αυτό είναι νομίζουμε μια μεγάλη επιτυχία το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανταποκρίθηκε στην πίεση ημών των σοσιαλδημοκρατών και άλλων για να υπάρχουν κεντρικά δημόσια αρχεία τα οποία θα περιέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για τους ε, πραγματικούς ε, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, τραστ, ε, ιδρυμάτων και διαφόρων τέτοιων κατασκευών. Τα μητρώα αυτά βεβαίως δεν είναι κάτι το αυτονόητο. Αυτό κατέστη σαφές στην αρχική πρόταση της Κομισιόν και τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο ήταν αντίθετα, όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε τελικά να επικρατήσει. Το τα μητρώ αυτά είναι υποχρεωτικά ε, τις ε, τράπεζες και στην διάθεση και όλων αυτών ε, των τραπεζών, των διοκτικών αρχών και των συμβολιογράφων και είναι στη διάθεση επίσης όσων θέλουν να αποδείξουν ότι είναι νόμιμα τα συμφέροντά τους αλλά και σε όσους κάνουν κάποια έρευνα για αυτά τα ζητήματα. Βεβαίως δεν θα πρέπει να έχουμε μεταβατικές περιόδους που ακούγονται για 4 ή 5 χρόνια και να εφαρμοστεί αμέσως και η διασυνοριακή πρόσβαση. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει η εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας και σε τρίτες χώρες. Έτσι θα μπορέσουμε πραγματικά να καταπολεμήσουμε το ξέβλημα χρήματος, ε, την φοροδιαφυγή και τις φορολογικές οάσεις. Όμως ε, το τελικό κείμενο προβλέπει πως ε, θα υπάρξει μια λίστα τρίτων χωρών στην οποία θα γίνεται σύγκριση και θα περιέχονται οι ελλείψεις τους σε σχέση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Απέναντι στις ε, προσπάθειες του Συμβουλίου, εμείς ως Κοινοβούλιο μπορούμε να ενημερώνουμε αυτόν τον κατάλογο μέσω πράξεων κατεξοδότηση κάθε τρεις μήνες. Εμείς θα θέλαμε κάποια πράγματα να πηγαίνουν ακόμη παραπέρα. Όμως σημειώνουμε πως ε, καταφέραμε να περάσουμε το βασικό μας αίτημα του Μητρώου αυτού. Αυτό μαζί με άλλες κατακτήσεις είναι μια επιτυχία της οδηγίας. Ε, παραμένουν όμως πάρα πολλά πράγματα άνοιχτα που πρέπει να γίνουν τα επόμενα πέντε χρόνια. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ. Επίτροπος κυρία Γιούροβα. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η έγκριση της τέταρτης αυτής οδηγίας και του σχετικού κανονισμού για την ενημέρωση για τη μεταφορά και τα χρημάτων και τα εμβάσματα θα αποτελέσουν ένα βασικό βήμα για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις προσπάθειες που κάνουμε ε, για να καταπολεμήσουμε την νομιμοποίηση των εισόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Θα ήθελα να εκφράσω την ε, τις μου προς ε, τους συνεισηγητές και το Κοινοβούλιο όπως επίσης και προς τους σκιώδεις ε, εισηγητές για την στεναρή του στήριξη προς τον κανονισμό αυτό και για τη σκληρή τους δουλειά. Επίσης, πολλές προεδρίες και κυρίως οι Ιταλικοί έκαναν πάρα πολλές προσπάθειες για να προωθήσουν το θέμα. Κάποια έκλεισαν το Δεκέμβριο πέρσι. Είμαι πεπισμένη πως σήμερα έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι ικανοποιητικό η αυριανή ψηφοφορία είναι ένα ακόμα βήμα έτσι ώστε να έχουμε πιο ισχυρούς κανόνες για να καταπολεμήσουμε την νομοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τροκρατρίας. Αυτά στα πλαίσια της ατζέντα για τα θέματα ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατόν τα εργαλεία αυτά, τα οποία μας επιτρέπουν καλύτερα να ανοιχνεύσουμε τα δις εκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες αυτές τις ροές του χρήματος που στηρίζουν τρομοκρατικές ομάδες και δράσεις. Έτσι ώστε να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι κάτοχοι λογαριασμών, κάτι το οποίο αποτελεί κομβικό σημείο ε, της ημερήσιας διάταξης σε επίπεδο και θα ήθελα να στηρίξω ε, κράτη-μέλη και του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου που ζήτησαν να δημιουργηθούν τα μητρώα των ιδιοκτητών των ε, εξωχώριων εταιριών. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως το πλαίσιο αυτό, το οποίο ε, εστιάζει στην αποτελεσματικότητα και στη μεγαλύτερη διαφάνεια, γρήγορα θα ε, μπει σε εφαρμογή. Πρέπει να επιταχύνουν τις προσπάθειες ε, εφαρμογή αυτών των απαιτήσεων τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να παροτρύνω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπερψηφίσει έτσι ώστε να έχουμε ένα πλαίσιο που θα μας επιτρέψει να καταπολεμήσουμε τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα ακολουθούν οι ομιλητές των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Ράντεφ για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το ξέβλημα χρήματος είναι 2,7% του παγκοσμίου ΑΕΠ, 1,6 τρισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, αλλά πραγματική, το πραγματικό κόστος είναι μεγαλύτερο, γιατί χρηματοδοτείται έτσι το οργανωμένο έγκλημα και η τρομοκρατία και αυτό επηρεάζει την ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο. Οπότε το τέταρτο πακέτο κατά του ξεβλήματος χρήματος είναι τόσο σημαντικό γιατί θα φέρει μεγαλύτερη διαφάνεια σε έναν όλο και πιο πολύπλοκο χρηματοοικονομικό κόσμο που αλλιώς θα είχε πολύ περισσότερες δυνατότητες για απάτη. Η συμφωνία για τους ε, τελικούς ε, δικαιούχους ε, της κάθε μαζί με τη συμφωνία για πιο αυστηρούς έλεγχους για τα εμβάσματα και τους ενδιάμεσους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών είναι σημαντικά στοιχεία στην νομοθεσία της Ένωσης. Έτσι θα έχουμε μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά την ιδιοκτησία εταιριών και μεγαλύτερη διαφάνεια στις ε, ε, εμπορικέ σχέσεις και θα λειτουργήσει καλύτερα η ενιαία αγορά. Ταυτόχρονα η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της νομοκρατίας θα διευκολυνθεί. Και αυτό είναι σημαντικό δεδομένης της τρομοκρατικής απειλής στην Ευρώπη. Και αυτή είναι μια νέα προτεραιότητα στην ε, Ευρωπαϊκή Ατζέντα της Ασφάλειας. Το τέταρτο πακέτο λοιπόν παρέχει επαρκή μέσα. Σας ευχαριστώ για δύο λεπτά κυρία Γκόμες. Με μικρόφωνο σας παρακαλώ. Is it working? Yes. Λειτουργεί. Ωραία ως ε, σκιώδης εισηγήτρια στην διαπραγματεύση της τέταρτης οδηγίας ε, για την ε, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητες πιστεύω ότι ε, γίνεται πιο ε, ε, σωστή η νομοθεσία και ευελπιστώ ότι θα ακολουθήσουν και οι χώρες. Βεβαίως η μεγαλύτερη καινοτομία είναι η ύπαρξη αυτού του νέου αρχείου που θα αποτελεί μητρό για όλες τις εταιρείε και για όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία. Πρέπει να πω πάντως ότι λυπούμε, είμαι απογοητευμένη γιατί παρά τον μεγάλο αριθμό οικονομικών σκανδάλων υστερεί η πρόταση της Επιτροπής σε διαφάνεια. Ε, εμείς είχαμε προβλέψει ως βουλευτές ένα ενιαίο σύστημα ε, και ενιαία φορολόγηση. Τώρα ε, υπάρχουν κάποια κενά όσον αφορά και την προσβασιμότητα του Μητρώου αυτού. Εν πάση περιπτώσει θα είναι 28 τα Μητρώα και 28 διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης. Επίσης παραμένουν και κάποια κάποιες ε, μορφές εταιριών έξω από το μητρό αυτό και επομένως χωρίς καμία προσβασιμότητα. Η δημιουργία αυτού του δημόσιου μητρώου μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Αυτό ενδιαφέρει ιδιαιτέρως ε, τους Ευρωπαίους πολίτες ε, οι οποίοι χυμάζονται από την εγκληματική οικονομική δραστηριότητα η οποία είχε ενταθεί και λόγω της κρίσης. Ωστόσο, δεν θα μας δώσει την δυνατότητα ε, να καταπολεμήσουμε αυτές τις αδιαφανείς δομές που χρησιμοποιούνται για την φοροαποφυγή. Θα πρέπει οπωσδήποτε να μεταφερθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα το νομοθετικό αυτό κείμενο έτσι ώστε να ε, αυξηθεί ε, η προσβασιμότητα σε όλες τις χώρες και έτσι ώστε να μπορέσουμε επιτέλους να δώσουμε ένα τέλος στους φιλολογικούς παραδείσους. Ευχαριστώ. Κύριε Γκόμες, δέχεστε μια ερώτηση από τον κύριο Σάνι. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ, αξιότιμα μέλη. Στις ε, παρεμβάσεις σας εστιάσατε σε μια σειρά από θέματα που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα επιβολής του κανονισμού και έχουμε το πρόβλημα τους φορολογικούς παραδείσους. Ρωτώ λοιπόν το εξής. Για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση και ολόκληρο το θεσμικό πλαίσιο δεν έχει ορίσει κάπου ε, τα, τους φορολογικούς παραδείσους. Ε, επειδή υπάρχει νομίζω άρνηση και έλλειψη βούλησης από τα κράτη-μέλη και την Κομισιόν για να αντιμετωπίσουν την άμεση ανάγκη για απόκτηση φορολογικών εσόδων, χωρίς τα οποία δεν υπάρχει υγιής ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά. Αυτή, αυτό ακριβώς προσπαθούμε να επιτύχουμε μέσω της Επιτροπής μας και είμαι σίγουρη πως εάν εμείς στο Κοινοβούλιο κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει θα μπορέσουμε να πείσουμε κυβερνήσεις και κομισιόν. Ευχαριστώ, κυρία Γκόμες. Η κυρία Φωνστόρχ, για ένα λεπτό. Ναι, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, μιλάμε σήμερα για βελτιωμένα μέτρα καταπολέμησης του ξεπλήματος ε, χρήματος ε, και όσα ε, υποκρύπτει η μαύρη εργασία, φοροδιαφυγή κτλ. Αλλά υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο εμφανίζεται, η κατάργηση των μετρητών συνολικά. Θα πρέπει να γίνουν όλες οι συναλλαγές ηλεκτρονικές για να είναι διαφανείς και να απαγορεύσουμε τα μετρητά. Ο Πέτερ Μπόφιγκερ, γερμανός ε, σοφός και ο επικεφαλής οικονομολόγος της Citibank στη Γερμανία το ζητάνε για άλλους λόγους αυτοί. Θα πρέπει λοιπόν οι υπάλληλοι να μπορούν να διαβάζουν κάθε μας συναλλαγή, πότε πίνω εγώ μια μπύρα και πότε παίρνω ταξί η ανωνυμία είναι προστασία των τρομοκρατών ή μήπως είναι και ένα θεμελιώδες δικαίωμα όλων των πολιτών. Δεν επιτρέπεται το να χάσουμε όλοι μας την ελευθερία μας ε, για να τιμωρηθούν μερικοί εγκληματίες. Σας ευχαριστώ για ένα μισή λεπτό, ο κύριος Τόρβαλτς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ξέρουμε, ε, το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος είναι ε, μεγάλο πρόσοδο, μεγάλη πρόσοδος για το ε, οργανωμένο έγκλημα και μεγάλη απώλεια πόρων για τις χώρες μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές, τους κοιόδης εισηγητές, όλοι δούλεψαν πάρα πολύ καλά για τα θέματα αυτά. Θα πρέπει πρώτα να δούμε τις αναλύσεις κινδύνου, risk analysis. Θα πρέπει αυτές οι αναλύσεις να είναι σωστές και επ' αυτόν να βασιστεί η δράση μας. Δηλαδή θα πρέπει πρώτα απ' όλα να μάθουμε ε, ποιος είναι ο πραγματικός ο, ε, ε, Θέλουμε μητρό πραγματικών ατόμων και πραγματικών νομίμων εταιριών. Αλλά περιπλέκεται το ζήτημα γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπως περιπτώσεις καζίνο με πολύ περίπλοκο ιδιοκτησιακό καθεστώς καθώς ε, και τελικά μπορεί να βρεθούμε απέναντι σε μια κατάσταση όπου αυτό που έχουμε δημιουργήσει ε, τελικά δεν ε, μας οδηγεί στο να πιάσουμε τους εγκληματίες γιατί αυτοί θα ξεφεύγουν, θα περνάνε μέσα από τους βρόχους του συστήματος. Θα πρέπει και σε κάθε χώρα να βελτιωθεί η νομοθεσία έτσι ώστε να λυθούν αυτά τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό η κυρία Καρή. Ε, ευχαριστώ. Ως ε, σκιώδης εισηγήτρια θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την εξαιρετική συνεργασία. Μπορούμε να πούμε ότι πετύχαμε πολλά. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Αν δούμε το τι συμβαίνει στον Παγκόσμιο Νότο, ο ΙΕ μας λέει πως οι χώρες Αφρικής χάνουν 50 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο λόγω φορολογικής απάτης και ξεπλήματος χρήματος. Τα διπλάσια σχεδόν από λαμβάνουν σε αναπτυξιακή βοήθεια. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει διαφάνεια. Είναι σημαντικό οι αρχές να μπορούν να διακρίνουν τι κρύβεται πίσω από τις διάφορες δομές που χρησιμοποιούν οι πολυεθνικές εταιρείε για να ξεπλύνουν τα χρήματα και να αποκρύψουν τα κέρδη τους. Και εργαστήκαμε πάρα πολύ σκληρά για να αποκτήσουμε ένα δημόσιο μητρό που θα καταστήσει δυνατόν να παρακολουθούμε τα ίχνη αυτών των εταιριών μέχρι τον πραγματικό ιδιοκτήτη. Αλλά όχι μόνο οι αρχές, οι απλοί πολίτες, οι και οι δημοσιογράφοι πρέπει να έχουν πρόσβαση γιατί εξάλλου χάρη στις δικές προσπάθειες είχαμε σκάνδαλα όπως το LuxLeaks. Δυστυχώς δεν ε, κατέστη δυνατόν να έχουμε ένα πλήρες ε, τέτοιο αρχείο γιατί οι ισχυρές δυνάμεις εντός της Κομισιόν και σε κάποιες χώρες εντός του Συμβουλίου δεν ήθελαν αυτή τη διαφάνεια. Απευθύνω λοιπόν έκκληση στις κυβερνήσεις μας και στην δική μου την κυβέρνηση της Δανίας να εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Ζολή για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Θα ήθελα να χαιρετήσω τις ε, σημαντικότατες ε, ε, προσπάθειες των εισηγητών και κυρίως την κυρία Σαρκεντίνη. Παρά τις σημαντικές πιέσεις θα έχουμε αύριο μητρό των εξωχωρικών εταιριών. Αυτό είναι κάτι σημαντικό, ένα μεγάλο και εκτιμένο. Όντως, μερικές χώρες έκαναν τα πάντα έτσι ώστε να ε, μειωθεί όσο γίνεται περισσότερο αυτή η πρόθεση. Ε, ε, θα πρέπει όμως να προσέχουμε κυρίως όσον αφορά τα τραστς και επίσης όσον αφορά την δυνατότητα πρόσβασης στα άλλα μητρώα των δημοσιογράφων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Εμείς πρέπει να να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας ε, να σταματήσουμε αυτές τις περίεργες διαδρομές των χρημάτων που τελικά ωφελούν τους τρομοκράτες, ε, τους ε, πλουσίους οι οποίοι δεν έχουν κανένα ηθικό φραγμό κλπ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φεράρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, στην Ευρώπη είναι χιλιάδες ε, οι οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις που έχουν πουλοκάμια ε, σε όλες τις χώρες και συνδέονται μεταξύ τους ε, όπως τα κινέζικα κουτιά. Ε, έγινε μια αξιολόγηση όσον αφορά το, ξέπλυμα, χρήμα, το ξέπλυμα χρημάτων και την σύνδεση με την χρηματοδότηση τρομοκρατίας ε, και, και ε, σημαντικό για να καταπολεμηθούν αυτές οι διαδικασίες είναι η συνεργασία. θα πρέπει όλα τα παράνομα φαινόμενα τα οποία αποτελούν παρέκκληση από την κανονική οικονομία θα πρέπει να, να καταπολεμηθούν. Θα πρέπει να αυξηθεί η χνηλασιμότητα των χρημάτων που μεταφέρονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ε, να ληφθούν τα μέτρα τα οποία θα κάνουν όσο γίνεται πιο διάφανες τις πράξεις και διαδικασίες των διαφόρων εταιριών. Να ξέρουμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης και ποιος έχει τη δυνατότητα λήψης ε, αποφάσεων. Ε, θα πρέπει να δίνεται δυνατότητα να συλλέγονται και να αποθηκεύονται σωστά αυτές οι πληροφορίες τις οποίες πρόσβαση θα πρέπει να έχουν όλοι. Ε, παρότι έχουμε πάρει κάποιες σωστές αποφάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν ατραπή, οι οποίες επιτρέπουν ε, στους εγκληματίες να ξεφεύγουν ε, και ε, να μην λησμονούμε ότι υπάρχουν και πολλές δυνατότητες που με επίσημο σχεδόν τρόπο μπορεί κανείς να φοροαποφύγει. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα σε αυτά τα στοιχεία γιατί διαφορετικά ε, θα έρεται η ίδια η αρχή της διαφάνειας. Ευχαριστώ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι σε αυτήν την έκθεση λείπει ή τουλάχιστον ακροθυγός αναφέρεται κάτι ε, το οποίο θα έπρεπε να βρίσκεται στο κέντρο των συζητήσεων, δηλαδή ε, τον κίνδυνο χρηματοδότησης μέσα από περίεργες οδούς ε, των Ισλαμικών ας πούμε οργανώσεων. Υπάρχει όμως μία ολόκληρη διασύνδεση ανάμεσα σε μαγαζιά που πουλάνε σε σφαγεία ή σε μουσουλμανικά, σε μαγαζιά που πουλάνε είναι μουσουλμανικά κρέατα, ε, τις ε, διάφορες θρησκευτικέ οργανώσεις. Υπάρχει μεγάλη διασύνδεση ανάμεσα σε αυτά ε, και γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει να κάνουμε μία κίνηση ευρύτερη από αυτήν που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και να λάβουμε υπόψη μας επομένως όχι για τις εγκληματικές οργανώσεις αλλά και τις τρομοκρατικές. Να αναρωτηθούμε, θέλουμε τελικά να δουλέψουμε σωστά έτσι ώστε να, να δούμε ποιος είναι αυτός ο οποίος ελέγχει αυτό το παράνομο, αυτή την παράνομη διαδρομή. Ευχαριστώ. Η κυρία Πάνοβα. Ευχαριστώ πολύ. Οι οικονομίες μας για να ευημερήσουν χρειαζόμαστε διαφάνεια και αξιοπιστία. Κάθε χρόνο στην Ευρώπη ο όγκος του χρήματος που παρανομοποιείται είναι διπλός από αυτά τα οποία έχουμε ε, τοποθετήσει στο πακέτο Juncker. Θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιούμε στην παιδεία, στην έρευνα, στην υγεία. Θα θέλαμε λοιπόν να είναι μεγαλύτερη η χνηλασιμότητα στα εμβάσματα έτσι ώστε να έχουμε περισσότερη ακαιρεότητα και να είναι πιο σταθερό και πιο αξιόπιστο το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα. Έχουμε λοιπόν τη δέουσα επιμέλεια και τα σχετικά εργαλεία. Να γνωρίζουμε τους πελάτες μας, να έχουμε καλύτερη κατανόηση του τι, ε, με τι ασχολούνται ε, οι πελάτες μας. Επίσης τα Μητρώα για το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης πραγματικός ιδιοκτήτης που θα κάνει το σύστημα πιο διάφανο και θα μας εμπιστεύεται περισσότερο πολίτης. Προστασία δεδομένων, ε, το θέμα αυτό σε σχέση με όσους βρίσκονται ε, στο Μητρό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί για την ε, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και για την νομιμοποίηση των εσόδων από δραστηριότητε. δραστηριότητες. Δεν μπορεί το θέμα αυτά να το αντιμετωπίσει ένα κράτος μέλος από μόνο του. Η νομοθεσία αυτή δημιουργεί πίστη στην αξιοπιστία του χρηματοπιστικού συστήματος, στο ότι χρησιμοποιούμε σωστά τα χρήματά μας και πίστη στο γεγονός πως η Ευρώπη θα ανακάμψει σε ένα δίκαιο περιβάλλον που θα βασίζεται σε νόμιμες πρακτικές. Ευχαριστώ για δύο λεπτά κυρία Φερέιρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τους εισηγητές, τους σκιώδες εισηγητές, τους συνεισηγητές για την τόσο ποιοτική δουλειά που έκαναν και καταλήξαμε σε μια συμφωνία υπό Ιταλική Προεδρία για ένα θέμα το οποίο είναι πολύ ουσιαστικό για να μην έχουμε φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή, απάτες και θα πρέπει το χρηματοπιστωτικό σύστημα να ενισχυθεί για να μπορεί να αντιμετωπίσει και την ονομοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και το θέμα της χρηματοδότησης τρομοκρατίας. Θα πρέπει λοιπόν να πετύχουμε το στόχο αυτό και να διώκονται όσοι κάνουν τέτοιες προσπάθειες στην Ευρώπη. Θα δημιουργήσουμε λοιπόν ένα ευρωπαϊκό μητρό για τους πραγματικούς ιδιοκτήτες ε, ή δικαιούχους αυτών των λογαριασμών ή εταιριών. Θα πρέπει να οργανωθούμε σε ευρωπαϊκό ε, επίπεδο για να δούμε ποια θα είναι η πρόσβαση σε αυτά τα μητρώα. Ο νόμος λέει πως χρειάζεται να αποδείξει κανείς το νόμιμο συμφέρον. Μα το νόμιμο συμφέρον πώς περιγράφεται. Γιατί τελικά είναι τα κράτη-μέλη τα οποία ενδεχομένως είναι λιγότερο απαιτητικά με τη διαφάνεια τη δυνατότητα να, να περιορίσουν την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες του Μητρώου. Επίσης, μπορούν να περιορίσουν τα κράτη-μέλη την πρόσβαση στα στοιχεία αυτά για περιπτώσεις τις οποίες χαρακτηρίζουν ως εξαιρετικές. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για ανήλικο ε, κάτοχο ή για κάποιον ο οποίος μπορεί να αποτελέσει θύμα εκβιασμού, απαγωγής, απάτης κτλ. Δηλαδή ε, ε, κάποιες περιπτώσεις οποίες είναι πολύ δύσκολο να ορίσουμε με σαφήνεια και εδώ απαγορεύουμε λοιπόν την πρόσβαση. Ε, βέβαια αποτελεί βελτίωση σε σχέση με τα όσα είχαμε στο παρελθόν. Είναι ένα πρώτο βήμα και νομίζω πως σε περιπτώσεις που δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε παραπάνω επριτάνευσε η ανάγκη του να υπογράψουμε ένα κείμενο το οποίο θα αποτελέσει μια βάση προσπάθειας. Ευχαριστώ πολύ. Φωτίκα. Κυρία Φωτίκα για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Μετά τις ε, επιθέσεις ε, στην Μαδρίτη, τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη δεσμεύτηκαν να καταπολεμήσουν την ε, τρομοκρατία και αυτό ισχύει και για τα δίκτυα της τρομοκρατίας. Δυστυχώς το επίπεδο της τρομοκρατικής απειλής δεν έχει πέσει όλα τα οικονομικά ή νομικά μέσα φαίνεται πως δεν επαρκούν. Γι' αυτό ακριβώς ε, η ευριανή ψηφοφορία έχει σχεδιαστεί για να καταπολεμήσει την τρομοκρατία και για μένα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους συντελεστές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γέζα και ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του ΕΛΚ για την στεναρή τους στάση στις διαπραγματεύσεις. Για εμένα η οδηγία υπογραμμίζει την σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην νομοθετική διαδικασία. Το ευρωπαϊκό αυτό μητρό τελικού δικαιούχου ήταν πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το υπερασπιστήκαμε στον τριμερή διάλογο. Η συμφωνία την οποία επιτύχαμε τον Δεκέμβριο ικανοποιεί το θεμητό αίτημα για μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση της καταπολέμησης του ξεπλήματος χρήματος. Υπάρχει όμως ακόμη πολύ μεγαλύτερο περιθώριο όταν μιλάμε για την προσβασιμότητα του αρχείου αυτού. Βεβαίω ε, υπάρχει και αυτή η έννοια του θεμητού συμφέροντο. Μετά την ψηφοφορία θα πρέπει να αναλάβουν τι ευθύνε του τα κράτη-μέλη και να κινηθούν γρήγορα για να εφαρμόσουν τους νέους ε, κανόνες ε, τα ενθαρρύνω να χρησιμοποιήσουν την ευελιξία που υπάρχει για να δώσουν απεριόριστη δημόσια πρόσβαση στα αρχεία αυτά για τους ε, δικαιούχους ε, εταιριών ε, και καταπιστευμάτων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, συνάδελφε. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Χρυσόγωνος. Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος αποτελεί μια τεράστια πληγή για την οικονομική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ελάχιστο άμεσο κόστος από το οργανωμένο έγκλημα ξεπερνάει τα 166 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της europol. αυτό σημαίνει λιγότερα χρήματα για την ανάπτυξη λιγότερα χρήματα για κοινωνικές παροχές και τελικά επίταση της κοινωνικής ανισότητας και αδικίας. γιατί όμως το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δεν έχει καταπολεμηθεί αποτελεσματικά ως τα σήμερα από το ευρωπαϊκό δίκαιο; η απάντηση είναι απλή διότι ποτέ ως σήμερα δεν υπήρξε η απαραίτητη πολιτική βούληση για αυτό εδώ έγκυται η χρησιμότητα των δύο νομοθετημάτων που συζητάμε σήμερα. φαίνεται πως επιτέλους κάτι αρχίζει να κινείται. οι προτάσεις από την ευρωπαϊκή επιτροπή έρχονται με βελτιώσεις σε σχέση με τα όσα ήδη ισχύουν. η τήρηση αρχείων με τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους ιδιοκτήτες των νομικών προσώπων συμπεριλαμβανομένων των καταπιστευμάτων που θα είναι ανοιχτά προς έλεγχο σε όσους αποδεικνύουν ένομο συμφέρον αποτελεί ένα πρώτο βήμα Προ την καθιέρωση ενό καθεστώτο διαφάνεια. χρειάζονται όμω και παραπέρα αποφασιστικά βήματα προ την κατοχύρωση τη διαφάνεια στι οικονομικέ συναλλαγέ. αυτή είναι η πραγματική και μεγάλη διαρθρωτική μεταρρύθμιση που χρειαζόμαστε και όχι η απορρίθμιση τη αγορά εργασία σε όφελο του κεφαλαίου την οποία προωθούν με κάθε τρόπο οι κυρίαρχε σήμερα στην ένωση πολιτικέ δυνάμει. Ευχαριστούμε κύριε Χρυσόγωνε. Κοράω για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ να σχολιάσω αυτό το τετάρτο πακέτο με τη σχετική νομοθεσία ε, για την ε, καταπολέμηση της νομοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελεί βήμα πρόοδου, παρόλο που ο δρόμος μπροστά μας είναι μακρύς. Για να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο, χρειαζόμαστε να κάνουμε πολλά βήματα ακόμα. Είναι μία από τις πληγές της εποχής μας, η οποία μας συμφέρει πολλούς. Είναι πολύ βολικό να έχεις πάντα κεφάλαια που να κυκλοφορούν στην αγορά, που είναι μάλλον άγνωστης προέλευσης, μάλλον από παράνομες δραστηριότητες, αλλά βολικό. Και υπάρχει και μια άλλη διάσταση, που καμιά φορά ξεχνιέται. Το γεγονός πως κάποια κράτη θα εφαρμόσουν μάλλον διαφορετικά αυτή την νομοθεσία. Κάποιοι θα τα πάνε καλύτερα σε επίπεδο εφαρμογής. Άρα λοιπόν είναι μια καλή ευκαιρία, αλλά θα πρέπει να συμμορφωθούν απόλυτα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, κύριος Μπριουά. Κύριε Πρόεδρε, Οποιαδήποτε ενίσχυση της νομοθεσίας χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας εκ των προτέρων θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό δεν θα πρέπει όμως να έχει ως επίπτωση την θυσία της λαϊκής κυριαρχίας και της κυριαρχίας των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία έχουν την ευθύνη να καταλημίσουν αυτές τις μαφίες. Θα πρέπει λοιπόν η νομοθεσία αυτή ε, να ακολουθεί από μια ενίσχυση της παρακολούθησης των κεφαλαίων που μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας μην είμαστε αφελείς. Η έλλειψη συνόρων χρησιμοποιείται από όσους προσπαθούν να ε, νομιμοποιήσουν παράνομα χρήμα κυκλοφορούν ελεύθερα τα κεφάλαια αυτά. Έχουμε ελεύθερη εγκατάσταση στα 27 κράτη-μέλη που έχει δημιουργήσει γόνιμο έδαφος σε αυτούς τους ε, εγκληματίες. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει αστυνομική συνεργασία, δικαστική συνεργασία αρκετά ισχυρή μεταξύ κρατών μελών, πιστεύω πως πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αναστείλουμε το Σέγγεν και τις ε, αρχές της ελεύθερης διακίνησης. Ο κύριος Μάνι, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάθε χρόνο έχουμε ένα ποσό μεταξύ 6,5 ε, δισεκατομμυρίων και 1,5-3 εκατομμυρίων που ξεπλένονται και αυτά με νόμιμους ε, τρόπους ε, όπως παραδείγματος χάρη τη κτλ. και τα λοιπά. Όλα αυτά επηρεάζουν τις ε, κοινωνίες μας ε, και την σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών ίδρυμάτων ε, και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στο σύστημα συνολικά. Οι διατάξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ακολουθούν τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις για να αντιδράσουμε αποτελεσματικά. Άρα χρειάζεται αυτό το αρχείο έτσι ώστε οι αρμόδιες αρχές να μπορούν να ξέρουν ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης των διαφόρων εταιριών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνει μια υπερεθνική αξιολόγηση κινδύνου και χρειάζεται άρα και μια εχνηλασιμότητα των εμβασμάτων. Διαφάνεια ναι, αλλά ταυτόχρονα σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Προστασία των προσωπικών δεδομένων. Προσωπικά δεδομένα δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται για επιχειρηματικούς σκοπούς. Η διεθνή συνεργασία λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική και θα πρέπει στοχευμένα να καταπολεμήσουμε το ξέπλυμα χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ευχαριστώ τον κύριο Κάρνης και τους άλλους εισηγητές. Ευχαριστώ κύριε Μάνα. Ακολουθεί ο κύριος Γκουαλτιέρη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θέλω ήθελα να πω ότι αυτή η δέσμη για το ξέπλυμα χρημάτων ε, είναι μια πολύ όμορφη σελίδα ε, στην κοινοβουλευτική ιστορία ε, και χαίρομαι γιατί έπαιξε σημαντικό ρόλο και συνέβαλε σε αυτό και η Ιταλική ε, προεδρία. Ε, εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτοι όσον αφορά τα διεθνή πρότυπα, ε, αλλά προχώρησε και παραπέρα το Κοινοβούλιο, βελτίωσε ακόμα περισσότερο τα πρότυπα. Δημιούργησε αυτή την ιδέα για το δημόσιο μητρό όσον αφορά τους υπεύθυνους των εταιριών και των ομίλων και επίσης σε σύνδεση με το άρθρο 30 αναφέρεται ότι ε, ε, νόμιμο συμφέρον δεν έχουν μονάχα αυτοί ε, που σχετίζονται με έσοδα από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση τρομοκρατίας αλλά και όλες οι κινήσεις εγκληματικών οργανώσεων που μπορεί να αφαιρέσουν χρήματα δημοσίου συμφέροντος. Και αυτό λοιπόν είναι μια ευρύτερη άποψη για την φοροδιαφυγή και για το οικονομικό θα συμφωνήσω με την εισηγήτρια ότι ε, αυτό είναι ένα μοντέλο στο οποίο θα πρέπει να ζητήσει η Ευρώπη από τους άλλους να προσαρμοστούν ε, και επομένως ε, θα πρέπει να επαγρυπνούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκαλτιέρη. Για ένα λεπτό ο κύριος Όζοκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι αυτή τη ε, στιγμή τα ζητήματα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του ξεπλήματος χρήματος είναι πάρα πολύ σημαντικά και χαίρομαι για το ότι λαμβάνουν υπόψη μια σειρά πτυχών και θεσμικών οργάνων που θα δράσουν σε αυτόν τον ε, τομέα. Θεωρώ πως πρέπει να ενισχύσουμε τους τομείς που αναφέρθηκαν δηλαδή πρώτα απ' όλα τις εγκληματικές δραστηριότητες ε, οι οποίες πράγματι αλλάζουν συνεχώς και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και βεβαίως να δράσουμε με τρόπο αναλογικό να λάβουμε επίσης υπόψη και τους παρόχους εμβασμάτων. Επίσης έχουμε και τις καταθυντήριες γραμμές ε, διεθνών οικονομικών οργανισμών με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφωθούμε. Σας ευχαριστώ για 1,5 λεπτό ο κύριος Βάλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ το Κοινοβούλιο που εργάστηκε με εξαιρετικό τρόπο. Ε, είναι προφανή τα βήματα προς τα εμπρός και πολυπληθή. Δυστυχώς ε, το Κοινοβούλιο πιεζόμενο από ε, ορισμένες ε, χώρες έκανε λίγο πιο, έβαλε λίγο νερό στο κρασί κάποιων προτάσεων. Η ύπαρξη ενός κεντρικού μήτρου όσον αφορά και τα καταπιστεύματα, όσον αφορά και τις εταιρείες με μονομένες ομίλους, τραστ κτλ. Ναι, ε, θα ήταν πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα κεντρικό και να είναι η πρόσβασή του ελεύθερη σε όλους. Ε, εν πάση περιπτώσει εδώ ε, για να έχει κανείς πρόσβαση θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει νόμιμο ενδιαφέρον. Επίσης τα περισσότερα τρας θα παραμείνουν εκτός του κεντρικού, εκτός των μητρώων και εν πάση περιπτώσει η πρόσβαση θα αφορά μονάχα αυτούς που κατέχουν ή ελέγχουν πάνω από το 25% ε, του μετοχικού κεφαλαίου και ενδεχομένως ε, ε, θα δημιουργηθούν επιπλέον προβλήματα. Σε εθνικό επίπεδο ενδεχομένως η εφαρμογή να γίνει με δυσανάλογο τρόπο στις διάφορες χώρες δημιουργώντας έτσι παραθυράκια και ατραπούς διεξόδου για πολλές εταιρείες. Το οργανωμένο έγκλημα ξέρουμε ότι κινείται και πολύ για τα πλοκάμια ότι είναι απλωμένα παντού. Ευχαριστώ, κύριε Βάλη. Ένα μισή λεπτό, κύριο Πέτερλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Παρόλη την νομισματική ένωση και την δημοσιονομική πολιτική πρέπει να καταπολεμήσουμε τις παράνομες ε, κινήσεις κεφαλαίων και συναριακέ μάλιστα. Καλώς ορίζω λοιπόν το ότι δεν είχαμε πολλές περιπλοκές ε, στις ε, συζητήσεις ε, τη στιγμή στην οποία συζητάμε την κοινή πολιτική ασφαλείας. Ξέρουμε λοιπόν πως οι παράνομες ροές συχνά καταλήγουν σε φορολογικούς παραδείσους. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ασκήσουμε πίεση στις χώρες που επιτρέπουν την ύπαρξη αυτών των Πρέπει λοιπόν να αυξήσουμε τη διαφάνεια, να συνεργαστούν μαζί μας και άρα είναι σημαντικό να εμπλέξουμε και τις υποψήφιες χώρες, οι οποίες θα πρέπει να σέβονται τις ίδιες προδιαγραφές και να προλαμβάνουν τις ε, παράνομες ροές. Το μισό λεπτό μου το αφήνω στον επόμενο μιλτή. Ευχαριστούμε. Για ένα λεπτό η κυρία Γιώτοβα. Три Είχαμε τρία νομοθετικά πακέτα τα οποία εγκρίθηκαν μέχρι στιγμή για να καταπολεμήσουν α, την νομιμοποίηση εισόδων από παράνομε δραστηριότητε. Δυστυχώ δεν ανταποκρίθηκαν στι προσδοκίε μα. Το έγκλημα πάντα είναι πιο ευέλικτο, πάντα είναι πιο γρήγορα από εμά. Χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται μια νέα πολιτική με δεσμευτικού κανόνε, με πολιτική δέσμευση να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα και θα πρέπει η Ευρώπη να ηγηθεί τη προσπάθεια να καταπολεμήσει του φορολογικού παράδεισου και α μην κλείνει τα μάτια. Παρακολουθεί τι επιδόσει τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι προσπάθειε που κάνουν να πατάξουν τη διαφθορά. Όμως η προσέγγιση αυτή έχει πια ξεπεράσει, έχει πια ξεπεραστεί, γιατί η έκθεση της κυρίας Μάλστρομ αποδεικνύει πως τέτοιου είδους προβλήματα έχουν όλες οι χώρες. Χρειαζόμαστε κοινή ευρωπαϊκή νομοθεσία, προσέγγιση της νομοθεσίας μας και του, ποινικού, και του συστήματος ποινικού δικαίου στα κράτη-μέλη και θα πρέπει η πολιτική αυτή να οδηγήσει σε νέες στρατηγικές για την ασφάλεια μέχρι το 2020. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φαντάλεν για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, το ξέπλυμα χρήματος ε, κοστίζει ε, κάθε χρόνο 1,5-3 εκατομμύρια ευρώ στην παγκοσμία οικονομία. Ένα τεράστιο ποσό που διακινούν ε, διακινητές ανθρώπων και ελαθρέμποροι ναρκωτικών. Η νέα λοιπόν αυτή νομοθεσία μπορεί να προσεγγίσει καλύτερα τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και το ξέπλυμα χρήματος και το στηρίζουμε. Και αυτό πραγματικά θα ωφελήσει τους ε, τίμιους συναλλασσόμενους οι οποίοι απλά τηρούν το νόμο. Ένα θέμα βεβαίως είναι ανησυχητικό η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Δεν θα πρέπει τα δεδομένα τα οποία είναι στη διάθεση των αρχών για αυτή και μόνο την υπόθεση να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς. Θα πρέπει να φροντίσουμε οι πολίτες και τα δεδομένα τους να είναι προστατευμένα. Ευχαριστώ κύριε Φαντάλεν. Η κυρία Μακοβέη για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Αγαπητή πολύ, κυρία Πρόεδρε. Το ξέπλυμα χρήματος. Να, κάνουμε επιτέλους ένα βήμα προς τα εμπρός. Για μια φορά θα καταφέρουμε να παρακολουθήσουμε τη διαδρομή του χρήματος γιατί θα πρέπει οι πολιτικές προσπάθειες που κάνουμε να βοηθήσουν να καταπολεμήσουμε τη χρηματοδότηση της ε, τρομοκρατίας. Τι σημαίνει αυτό το μητρό, ότι μας δίνουν τα πραγματικά στοιχεία των ιδιοκτητών, των δικαιούχων αυτών των λογαριασμών και πολλές φορές ε, οι δημοσιογράφοι μόνο μπορούν να αποδείξουν ε, τα στοιχεία αυτά γιατί εμείς πώς αποδεικνύουμε το νόμιμο ε, συμφέρον όταν υπάρχει πραγματικό εμπόδιο στο να έχουμε πρόσβαση στα μήτρο αυτά. Έχουμε κάποιες εταιρείε φαντάσματα οι οποίες με την οδηγία αυτή δεν πρόκειται να αποκαλυφθούν. Έχουμε πολυεθνικές οι οποίες κερδίζουν τεράστια ποσά και τα μεταφέρουν σε φορολογικούς παραδείσους. Το κέρδος πάντα ε, αποτελεί τον απότερο στόχο όλων αυτών και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνουμε αυτό το θέμα. Έχουμε φορολογικού παραδείσους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Λουξεμβούργο, δισεκατομμύρια που έχουν χαθεί σε φόρους από τους πολίτες μας γιατί βεβαίω οι επιχειρήσει αυτέ δεν πληρώνουν φόρους όπως θα έπρεπε. Επίσης τα καζίνο ξεπλένουν χρήμα κάθε βράδυ. Στην Ήπειρό μας δεν υπάρχει ε, υποχρέωση να ξέρει κανείς ποιοι είναι οι πελάτες του. Για μια φορά ακόμα λοιπόν θα πρέπει να απευθύνω μια έκκληση. Ευχαριστώ για ένα λεπτό η κυρία Σλάιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τις προσπάθειες ε, που κατέβαλαν, ευχαριστώ τους συνάδελφους για τις ε, προσπάθειες που κατέβαλαν. Σημαντικό βήμα κάνει η Ευρώπη όσον αφορά το ξέπλυμα ε, χρήματος και τη χρηματοδότηση της δημοκρατίας, οργανωμένο έγκλημα κτλ. Το Μητρό καταγραφής πλέον είναι υποχρεωτικό και εκεί θα καταγράφονται υποχρεωτικώς όλα τα ιδιοκτησιακά καθεστώτα των εταιριών και των τραστ. Βεβαίως θα έπρεπε να είμαστε πιο θαραλέοι Βεβαίω Βεβαίως θα έπρεπε να έχει πρόσβαση και κάποιος στα μητρώα αυτά, κάποιος που δεν μπορεί να αποδείξει το νόμιμο ενδιαφέρον. Η διαφάνεια είναι θεμελιώδους σημασίας. 70% των περιπτώσεων παράνομη διακίνησης χρήματος αφορά από ό,τι φαίνεται εταιρείε φαντάσματα. Ε, όλα αυτά κοστίζουν εκατομμύρια και στον αναπτυγμένο κόσμο αλλά κυρίως στον αναπτυσσόμενο. Ελπίζουμε ότι η οδηγία αυτή θα αποτελέσει στο πρώτο βήμα μιας μακράς οδού και διαδικασίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό ο κύριος Βιασντόφσκι. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Εγώ είμαι επιφυλακτικός γενικά, αλλά δεν έχω καμία αμφιβολία πως ε, θα πρέπει να είναι αυστηροί οι κανόνες όταν μιλάμε για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε για τέτοια μέσα. Είμαι ικανοποιημένο ε, με το μητρό αυτό, αλλά δεν συμφωνώ πως θα είναι κατά τη ιδιωτικής ζωή των πολιτών. Ας μην διστάζουμε. Θα μας βοηθήσει να καταπολεμήσουμε, νομίζω, τη ξέπλυμα χρήματος. Και τέλος θα πρέπει να εφαρμοστεί με τρόπο σωστό. Κάποια πράγματα δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί. Ευχαριστώ. Η κυρία Πιτέρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ξέπλυμα χρήματος συνδέεται άμεσα με το οργανωμένο έγκλημα και αυτό επηρεάζει ιδιαίτερος την διεθνή οικονομία. Ε, το FATF ε, ε, κατέδειξε σαφώς ότι μιλάμε για 2,7% του παγκόσμιου ΑΕΠ με αυξητική τάση χρόνο με το χρόνο. Η τεχνολογική πρόοδος βεβαίως, ε, ε, η ελεύθερη κυκλοφορία ε, των κεφαλαίων, τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν σε όλη αυτή την διαδικασία. Και αν προσθέσουμε και το τραπεζικό απόρριτο, είναι εύκολο τελικά να κρύψει κανείς ε, ε, έσοδα ε, και με την ίδια ευκολία μπορεί να χρηματοδοτήσει εγκληματικές δράσεις ή τρομοκρατία. Γι' αυτό λοιπόν το μητρό το οποίο ε, προτείνεται είναι πολύ σημαντικό. Θα μας βοηθήσει οπωσδήποτε ε, να ε, χτυπήσουμε την χρηματοδότηση της διεθνούς τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Ελπίζουμε ότι θα καταπολεμήσουμε με τον τρόπο αυτό αυτές τις πληγές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Στεχόφσκι για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί εισηγητές, να σας ευχαριστήσω θέρμα για τη δουλειά που έχετε κάνει στην οδηγία αυτή. Είμαι υπερήφανος ε, για το ότι η Τσέχα Επιτροπός έφερε αυτό το έγγραφο. Πραγματικά βοηθάει την Ευρώπη να προχωρήσει στην καταπολέμηση παράνομων δραστηριοτήτων απάτης και εξεπλήματος χρήματος. Και τα ποσά που αναφέρονται είναι πράγματι ανησυχητικά. Κανείς μας δεν μπορεί να πει από πού ξεκινάνε και πού πάνε τα λεφτά και ποιον ωφελούν. Άρα είναι απολύτως απαραίτητο να παρακολουθούμε αυτές τις συναλλαγές μακροπρόθεσμα και με διαφάνεια. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ μιας οικονομίας χωρίς μετρητά. Μια τέτοια οικονομία θα προχωρήσει την Ευρώπη πιο μακριά στην καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος. Να τονίσω και κάτι άλλο που δεν άκουσα. Μια άλλη πτυχή αυτών των δραστηριοτήτων είναι ότι είναι διεθνείς ε, και ε, ακολουθούν αναπάντεχες κατευθύνσεις. Δεν πρέπει λοιπόν να περιοριστούμε εντός της Ένωσης, αλλά να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας σε διεθνές επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στη διαδικασία και Η κυρία Γκάλ Πέλτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Σήμερα το ξέβλημα χρήματος είναι ένας πάρα πολύ επικερδής ε, κλάδος ε, και βεβαίως έχουμε συνεχώς νέες διατάξεις αλλά δεν ξέρουμε τι κάνουν οι εγκληματικές ε, οργανώσεις. Εγώ συμφωνώ όταν λέμε πως ε, θα πρέπει να εκπληρώνουν τις διατάξεις και υποκείμενα λοδαπού δικαίου όταν μιλάμε για ζητήματα διαφάνειας. Θα πρέπει να βελτιωθούν νομίζω τα αρχεία αυτά, θα πρέπει να έχουμε πληροφορίες για τον τελικό δικαιούχο. Δεν είναι πάρα πολύ απλό αυτό. Θεωρώ πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλή δουλειά να κάνει ακόμα, αλλά έχουμε ένα καλό μέσο. Σας ευχαριστούμε. Η ε, κυρία Φρουντσουλίκα έχει το λόγο. Μεγάλη χαρά. για μας. Μεγάλη χαρά να μας δίνετε το λόγο εσείς. Come Μ' αρέσει που έχουμε συμπεριλάβει εδώ αυτή τη δυνατότητα να έχουμε ένα μητρό κατόχων ε, και ειδικά ε, την ε, διατύπωση που λέει νόμιμο συμφέρον και ικανή πρόσβαση. Έτσι τα κράτη-μέλη που το επιθυμούν μπορούν να δώσουν ένα πιο διευρυμένο ορισμό του τι σημαίνει νόμιμο συμφέρον. Θα μπορούσε αυτές οι πληροφορίες να είναι ανοιχτές κατά περίπτωση και βέβαια υπό εξαιρετικές ε, συνθήκες εάν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος βίας, εκβιασμού, απαγωγής κτλ ή σε περίπτωση που είναι ανήλικος ή ε, κτλ. Στην περίπτωση αυτή νομίζω πως θα έχουμε τη μέγιστη διαφάνεια και αυτό θα μας εξηγεί σε κάθε περίπτωση ποια είναι η κατοχή των ε, εταιρικών αυτών σχημάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγμα το οποίο είναι θαυμάσιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα έχει το λόγο στα πλαίσια του Catch the Eye. Ο επόμενος ομιλητής, παρόλο που εσείς δεν είσαστε πάντοτε παράδειγμα συμπεριφοράς, επόμενη... Οι αλλαγές έδωσαν την ευκαιρία στις πολυεθνικές να φοροδιαφεύγουν, διότι δεν φορολογούνται εκεί όπου παράγονται τα κέρδη, αλλά σε φορολογικούς παραδείσους και αυτό σημαίνει απώλεια δισεκατομμυρίων ευρώ από τις χώρες της αφρικής από τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου. ταυτόχρονα πολλές μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελλάδα φοροδιαφεύγουν έχοντας εγκατασταθεί φορολογικά είτε στην ολλανδία είτε στο λουξεμβούργο όπου είχαμε και το γνωστό σκάνδαλο των luxleaks. πρέπει επίσης να χτυπηθεί η πρακτική των offshore εταιριών που συμβάλλουν στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος τέλος πρέπει να ληφθούν μέτρα για να καταπολεμηθούν οι τζιχαντιστές που χρηματοδοτούνται με την πώληση πετρελαίου στις χώρες της δύσης. για τον λόγο αυτό συμφωνούμε με την τήρηση κεντρικών δημοσίων αρχείων για τους πραγματικούς ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων. πρέπει όμως να υπάρξουν εγγυήσεις για την χρήση των προσωπικών δεδομένων. διαφωνούμε όμως με την εξαίρεση των καζίνο και των τυχερών παιχνιδιών από την εφαρμογή της νομοθεσίας. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μαριά. Ο κύριος Γιάκοφιτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύρια Επιτροπέ, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί εισηγητές, θα ήθελα ε, να καλωσορίσω αυτό, αυτή τη νέα ε, πρόταση και να πω ότι αποτελεί ένα εξαιρετικό βήμα προς τα εμπρός. Αλλά ένα βήμα μόνο ε, ε, που θα πρέπει να ενθαρρυνθεί έτσι ώστε να προχωρήσουμε αν πραγματικά θέλουμε να καταπολεμήσουμε αυτό το ξέπλυμα ε, του χρήματος που διαρκώς παίρνει χρήματα από την οικονομία μας. Υπάρχουν δύο προβλήματα. Πρώτα απ' όλα ότι ε, όλα θα εξαρτηθούν από την βούληση των κρατών μελών να καταπολεμήσουν την νομοποίηση των εισόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Θα πρέπει να είμαστε ε, σαφείς και καθαροί. Δεν είναι δυνατόν να λύσουμε τα προβλήματα αυτά εάν δεν συνεργαστούμε στενά με τις τρίτες χώρες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιάκοφτσίτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και η οδηγία και ο κανονισμός ε, πάνε προς, τον, ε, ε, προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά δεν χρειάζεται να πανηγυρίζουμε γιατί εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλη απειλή για τα οικονομικά μας συστήματα η νομιμοποίηση εισόδων από παράνομες δραστηριότητες, η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή. Εκατομμύρια ζημιά κοστίζει κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι επιλογές δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές. Ευελπιστώ ότι θα συνεχίσουμε αυτό το πρώτο βήμα προς την καλή κατεύθυνση. Όσον αφορά ε, το Μητρό των Ιδιοκτητών, αυτό ήταν ένα πραγματικά μεγάλο βήμα προς ε, την κατεύθυνση της ε, διαφάνειας. Ξέρουμε ότι δεν είναι πάντα εύκολο να βρει κανείς ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, αλλά ξέρουμε ότι αυτό το ξέπλυμα χρήματος είναι μια μεγάλη πρόκληση για όλους μας και για όλες τις οικονομίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σόλτες. Τελευταίος ο κύριος Σβέρ στη διαδικασία και έτσι Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ τους εισηγητές για τη δουλειά που έκαναν. Ακούσαμε ήδη πως η παγκόσμια οικονομία χάνει γύρω στο 5% του ΑΕΠ και βεβαίω αυτό επηρεάζει τη φτώχεια. Φαντάζεστε μια κατάσταση στην οποία όλα αυτά τα λεφτά θα πήγαιναν να, ε, να επενδυθούν σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε αποτελεσματικότερα μέτρα από την αστυνομία, τις φορολογικές αρχές, τις διοκτικές αρχές, καλύτερα αρχεία των ε, δικαιούχων και βεβαίως ε, καλύτερη παρακολούθηση των φορολογικών παραδείσων και βεβαίως τα παγκόσμια προβλήματα απαιτούν πάντα μια ολιστική προσέγγιση θεωρώ πως είμαστε σε καλό δρόμο και θα αντιμετωπίσουμε καλύτερα το οργανωμένο έγκλημα. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο έχει η κυρία Επίτροπος. Ευχαριστώ πολύ. Η συζήτηση η οποία μόλις έγινε με εντυπωσίασε και ελπίζω πως η αδριανή ψηφοφορία θα μας βοηθήσει κάτι να πετύχουμε. Τα θετικά αποτελέσματα τα οποία μόλις περιγράψαμε και τα οποία καλό θα ήταν ε, να επιδιώξουμε μέσω αυτών των δύο κειμένων. Σας άκουσα. Μιλήσατε πολύ για το ποινικό δίκαιο, για την προστασία των δεδομένων. Θα ήθελα να σας δώσω και εδώ κάποια στοιχεία για το πώς μπορούμε να ασχοληθούμε με το θέμα του οργανωμένου εγκλήματος. Να σας πω πως ε, αντιμετωπίζουμε το θέμα σφαιρικά. Για να πατάξουμε το έγκλημα και στο χώρο του ποινικού δικαίου εμείς ενισχύουμε τη συνεργασία μεταξύ της Eurojust και της Europol με εμάς ε, κυρίως για να έχουμε ένα καλύτερο επίπεδο ασφάλειας στην Ευρώπη και για τις τρεις τρίτες χώρες στις οποίες αναφερθήκατε και την ανάγκη που έχουμε να διευρύνουμε εκεί τις δράσεις μας και να δούμε τι θα γίνει με τους υπηκόους τρίτους χωρών. Να σας πληροφορήσω πως στα πλαίσια του θεματολογίου για την ασφάλεια έχουμε ως σκοπό ε, το Μητρό ε, ε, Εγκληματιών Υπηκών Τρίτων Χωρών να το ενισχύσουμε έτσι ώστε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για τις ε, ροές υπόπτων ε, και αυτούργων. Μιλήσατε για προστασία δεδομένων και με μεγάλη ικανοποίηση αναγνωρίζω πως είμαι υπεύθυνη και για αυτόν τον κανονισμό γιατί η προστασία των δεδομένων είναι μια μεταρρύθμιση την οποία τώρα ε, κλείνουμε, φέτος ελπίζω στο Συμβούλιο Θα γίνει και τριμερής διάλογος την επόμενη χρονιά και αποτελεί πραγματική επανάσταση γιατί θα, αντικαταστήσει τα 23 εθνικά συστήματα με ένα πανευρωπαϊκό σύστημα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μιλώντας λοιπόν για προστασία δεδομένων σε σχέση με την οδηγία για το ξεπλήμα χρήματος, να σας πω πως δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και κυρίως στο δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και στην προστασία των ε, προσωπικών στοιχείων. Αυτά λοιπόν τα νομοθετικά κείμενα είναι πολύ συμβατά μεταξύ τους και νομίζω θα συνδυαστούν πολύ καλά και στην πράξη. Για το πακέτο αυτό με ικανοποίηση άκουσα πως θεωρείται πως είναι λογικό, ευχριστό, απαραίτητο, αναλογικό και θα αποτελέσει του, τη βάση για να καταπολεμήσουμε το έγκλημα στην οικονομική ζωή της Ευρώπης. Όχι μόνο καταπολέμηση λοιπόν του οργανωμένου εγκλήματος, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα και άλλα σχετικά αδικήματα, αλλά παράλληλα και αυτό που αναφέρατε σε πολλές φορές, πολλές φορές οι συνάδελφοι εδώ, η τρομοκρατία όχι μόνο για να εξοικονομήσουμε χρήματα, και να μην εξαφανίζονται τα χρήματα αυτά, αλλά για να χρησιμοποιούνται καλύτερα. Το είπατε συχνά. Δεν είναι όμως μόνο θέμα εξοικονόμησης, αλλά είναι και θέμα προστασίας ανθρώπινης ζωής γιατί οι οικονομικές αυτές συναλλαγές πολύ συχνά αποτελούν τα πρώτα μηνύματα πως υπήκεται μια τρομοκρατική δραστηριότητα ή επίθεση. Άρα λοιπόν είναι ουσιαστικό να μπορούμε να παρακολουθήσουμε το σημείο αυτό για να ισχύσουμε τα επίπεδα ασφάλειας στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ και πάλι για τη στήριξη που προσφέρατε και ελπίζω πως αύριο η ψηφοφορία θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ comisar, rog pe domnul Carins ia cuvântul Ο κύριος Κάρινς για δύο λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα για μία ακόμα φορά να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την συνεργασία τους στην προετοιμασία αυτής της έκθεσης. και ξέρουμε πλέον ότι από όλε τι ομάδες υπάρχει μια καλή στάση έτσι ώστε ε, να προχωρήσουμε στην δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μητρώου και να καταπολεμήσουμε τελικά ε, αυτή την ε, πληγή που είναι το ξέπλυμα χρήματος. Ευχαριστώ η κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλοί από τους συναδέλφους μου είπαν ότι το δημόσιο μητρό δεν θα είναι πραγματικά δημόσιο γιατί θα πρέπει να αποδείξεις ότι έχεις νόμιμο ενδιαφέρον για να το συμβουλευτείς. Πάντως πρέπει να πω ότι αναφέρεται ότι η αρχή ε, θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν έχει κανείς ένομο ε, ε, συμφέρον. Ε, και ότι μπορεί να φτάσει και μέχρι το, τα δικαστήρια ε, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει εάν κάποιος έχει ή όχι ένομο συμφέρον και αν φτάσουμε μερικές φορές στα δικαστήρια νομίζω ότι ε, εύκολο, εύκολο θα είναι πλέον να αυξηθεί αυτή η προσβασιμότητα γιατί δύσκολο ένα δικαστήριο θα πει σε έναν πολίτη ότι δεν έχεις ένομο συμφέρον να ε, έχεις πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες οι οποίες αφορούν ε, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος ε, κτλ. Εάν εμείς εδώ αποφασίσουμε ότι πραγματικά θέλουμε να προχωρήσουμε τότε θα ανοίξουμε σιγά σιγά τις διόδους έτσι ώστε να είναι πραγματικά δημόσιο αυτό το Μητρό. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση και ευχαριστώ και την ε, κυρία Επίτροπο για τα σχόλια τα οποία έκανε. Θα ήθελα ε, να πω ε, ότι εγώ ε, ε, προσπάθησα να βελτιώσω την τέταρτη οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος και τις μεταφορές χρηματικών ποσών. Υπάρχει ένα ζήτημα όσον αφορά τις, τα προσωπικά δεδομένα τα οποία πραγματικά αφορούν συγκεκριμένα άτομα και επομένως θα πρέπει η προστασία να είναι εξασφαλισμένη. Ε, ξέρουμε ότι χρησιμοποιούν οι εγκληματίες και οι εγκληματικές οργανώσεις ένα σωρό τεχνικά τερτύπια και όλες τις προόδους της τεχνολογίας έτσι ώστε ε, να ξεφύγουν. Ε, θα πρέπει να το δούμε, θα πρέπει να βρούμε λύσεις οι οποίες να λειτουργούν και να πω επίσης ότι ευχαριστώ όλους όσοι συνεργάστηκαν έτσι ώστε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πέτερ ναι, κύριε Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την συνεργασία και να πω πως ε, σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι με το κεντρικό αυτό αρχείο για να υπάρχει μια διαφάνεια. Θα πρέπει όμως επίσης να είναι σαφές ότι η καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος και της απάτης είναι συνεχής γιατί οι μέθοδοι εξελίσσονται συνεχώς. Οπότε θα πρέπει και εμείς μετά την αυριανή ψηφοφορία να μπορούμε να αντιδρούμε και να είμαστε ακόμη πιο φλόδοξοι. Γι' αυτό ο συμβιβασμός με το Συμβούλιο είναι άλλο ένα νέο βήμα, που όμως πρέπει να συνεχιστεί. Πρέπει να υπαγρυπνούμε να εφαρμοστούν αποτελεσματικά αυτές οι διατάξεις και ειδικά τα κράτη-μέλη να επιτρέψουν ε, την πρόσβαση σε αυτό το αρχείο σε άτομα με θεμητά και ένομα συμφέροντα. Επίσης θα πρέπει να διευκολυνθεί η διασυνοριακή πρόσβαση. Δεν καταλαβαίνω γιατί χρειάζεται τέσσερα χρόνια για την διασύνδεση των εθνικών αρχείων όταν θεωρητικά είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες. Θεωρώ λοιπόν πως όλοι εδώ πέρα πρέπει να καταβάλουμε μια κοινή προσπάθεια γιατί η προσπάθεια αυτή δεν γνωρίζει σύνορα, πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Σας ε, ευχαριστώ. Θα ψηφίσουμε λοιπόν αύριο, λίγη προς το παρόν εδώ η συζήτηση. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για μια κοινή συζήτηση που θα γίνει για τις διαδικασίες αφαιρεγγιότητας. Έχουμε εδώ μια σύσταση σε δεύτερη ανάγνωση. Ο κύριος Ζήφ